So, uh, uh, ήρθατε στην ε, δέκατη Σύνοδο ΑΣΕΠ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια οργανωτικά και κατόπιν θα περάσουμε στην έναρξη της συνεδρίασής μας. Είμαι συμπρόεδρος από την ευρωπαϊκή πλευρά εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και οι δύο συμπρόεδροι κάθονται δίπλα μου η κυρία Σάιτουρη που είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Μπαγκλαντές και ο κύριος Ράιεν ο πρόεδρος της Γερουσίας της Αυστραλίας. Θα ήθελα να ανακοινώσω ότι πέρα από τις συνήθεις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε ρωσικά στο κανάλι 27 σε μέρες, στο 25 και σε βιετναμέζικα στο κανάλι 26 και μογγολικά στο κανάλι 29. Έχουμε ένα μεγάλο εύρος γλωσσών σήμερα. Έχουμε προγραμματίσει τέσσερις δηλώσεις κατά την έναρξη της συνεδρίασης και θα σας ζητήσω να περιοριστείτε στα 10 λεπτά καθώς δεν έχουμε πολύ χρόνο. Καταρχήν, ε, της αρχής δεν ε, θα ανοίξουμε τη συζήτηση εκτός και αν έχει απομείνει κάποιος χρόνος. Αυτό εξαρτάται από τις εισαγωγικέ ομιλίες, αλλά αργότερα στα πάνελ ελπίζω ότι θα έχουμε ιδιαίτερα Ενδιαφέρουσε και έντονες συζητήσει και ιδιαίτερα αύριο στην Ολομέλεια. Και θα ήθελα να σημειώσετε ότι μόνο τα μέλη των κοινοβουλίων καλούνται να πάρουν το λόγο. Μία κοινή δήλωση είναι υπό εκπόνηση στην Συντακτική Επιτροπή. Ήδη σήμερα το πρωί κάναμε αρκετή δουλειά σε ένα πολύ καλό πνεύμα. Και... Αργότερα θα έχουμε το τελικό κείμενο που θα υιοθετηθεί αύριο στα τέλη της ε, διαδικασίας ακριβώς πριν τις 12 πριν από την καταληκτήρια συνεδρίαση ε, θα μεταδίδονται ζωντανά οι συζητήσεις μας ε, και από την τηλεόραση του Κοινοβουλίου, η PTV, επομένως μπορούν και οι συνάδελφοι στις εκλογικές τους περιφέρειες ε, να σας παρακολουθήσουν. Και μετά την ε, πρωινή συνεδρίαση θα έχουμε και μια οικογενειακή φωτογραφία. Θέλω να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο της Μογγολίας ε, που φιλοξένησε την ΑΣΕΠΕΝΙΑ στο Ουλάν Μπατόρ το 2016. Η συνεδρίαση εκείνη, η συνοδος εκείνη ήταν πολύ επιτυχή στο Ουλάν Μπατόρ και θα ήθελα τώρα να σας ε, καλωσορίσω εκ μέρους του κυρίου Ταγιάννη, του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τα θέματα που αποφασίσαμε να σας παρουσιάσουμε για συζήτηση και για εξαγωγή συμπερασμάτων κατά την ΑΣΕΠ 10. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά μας να καλωσορίσουμε τις πολυάριθμες αντιπροσωπείες από την Ασία και την Ευρώπη σε αυτή την ε, δέκατη κοινοβουλευτική διάσκεψη Ασίας-Ευρώπης. Και ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε τόσο πολλοί αριθμούς ε, εκπροσώπους ε, ε, των κοινοβουλίων είναι η πρώτη φορά που το κοινοβούλιο έχει το προνόμιο να φιλοξενεί τόσο σημαντική συνάντηση. Χαιρόμαστε να σας καλωσορίζουμε στις Βρυξέλλες και σε αυτό τον Νίκο πρόκειται για ένα φανταστικό υπερεθνικό κοινοβούλιο ε, που εκπροσωπεί πάνω από 500 εκατομμύρια πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την συμμετοχή των πολιτών. Επίσης, χαίρομαι να καλωσορίσω τον πρόσωπο της ε, Μογγολίας που μας ε, φιλοξένησε το 2016 και πάλι έχω την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω για μια πολύ επιτυχή συνάντηση. Φέτος ε, το κύριο θέμα επικεντρώνεται στον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής σε διάφορους τομείς της ζωής και δεν θα μπορούσε παρά να είναι ιδιαίτερα επίκαιρο. Πάρα πολλοί από εμά έχουμε βιώσει τα δεινά που υφίστανται οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, ακόμη και στη Φιλανδία, στη χώρα μου. Είχαμε ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι. Εγώ προσωπικά δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η χώρα μας ε, που είναι ε, ε, τόσο πλούσια ε, σε υδάτινους σπόρους ε, είχε τόσο μεγάλη ξηρασία και είχαμε επιπτώσεις στη γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα στον κατάλογο των ακραίων καιρικών φαινομένων που βιώνουμε. Πιστεύω ω βουλευτές από την Ευρώπη και την Ασία έχουμε πολλά να πετύχουμε προκειμένου να μπορέσουμε ε, να έχουμε φιλόδοξους ε, στόχους για το κλίμα στα πλαίσια τη Συνόδου των Παρισίων. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για το 2030 με τους 25 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο για μας για να το εφαρμόσουμε. και περί φιλοδοξίας και εφαρμογής. Και θα ήθελα να πω ότι ουσιαστικά σε αυτή την ε, νέα ατζέντα έχουμε ε, μία πρόκληση για τη λήψη αποφάσεων. Θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη διαδικασία λήψης αποφάσεων για να αντιμετωπίσουμε ταυτόχρονα πολλαπλές προκλήσεις. Γιατί αν προσπαθήσουμε να λύσουμε ένα μονοθέμα μπορεί να δημιουργήσουμε ένα άλλο πρόβλημα. Σε όλες τις δράσεις για το κλίμα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι σεβόμαστε τα δικαιώματα των αυτόχθονων λαών και τα δικαιώματά του στη γη βλέπουμε μερικές φορές διάφορα παζαρέματα και θέλουμε να αποφύγουμε τέτοια παζαρέματα και όσο είναι δυνατόν. Εμείς ανυπομονούμε να μοιραστούμε τις εμπειρίες μας, τις βέλτιες πρακτικές ε, και να ακούσουμε και τις ε, ε, δικές σας εμπειρίες καθώς κάποιοι εταίροι από την Ασία είναι στην πρώτη γραμμή τη καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και ίσως και εκεί να είναι σε ηγετική θέση στο να ε, υιοθετήσουν ε, τα ηλεκτρικά οχήματα και να μεταμορφώσουν ε, τα συστήματα κυκλοφορίας. Όλοι πρέπει να επιταχύνουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ξέρουμε ότι στην Ασία κάποιες από τις πιο ευπαθείς ομάδες πραγματικά υποφέρουν και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στην κατάσταση των πιο ευάλωτων ανθρώπων, των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες, στις γυναίκες, στους εκτοπισμένους. Κάποιοι που εκτοπίστηκαν και λόγω της κλιματικής αλλαγής. Αυτό πρέπει να είναι μέρος της δράσης μας για το κλίμα. Ο διάλογο και η συνεργασία με τα χρόνια μεταξύ Ευρώπη και εσείς έχουν αυξηθεί, έχει αυξηθεί σημαντικά και είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπουμε πόσο ενεργή έχει γίνει η διαδικασία ΑΣΕΜ και την υποστηρίζουμε Εμεί, οι βουλευτέ, έχουμε σημαντική συνεισφορά στη διαδικασία. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε πώ θα ενδυναμώσουμε την κοινοβουλευτική διάσταση τη διαδικασία του Ουλάν Μπατόρ και ευχαριστώ ε, τους ε, υποδε που μας φιλοξένησαν. Πώς μπορούμε να έχουμε ένα πιο μόνιμο διάλογο και επικοινωνία μεταξύ μας προκειμένου να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας, οι λαοί μας και ο πλανήτης μας σήμερα. Κατά την άποψή μου, και εδώ μιλώ εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν αρκεί να θετούμε μια κοινή δήλωση, μια κοινή διακήρυξη κάθε δύο χρόνια. Δεν αρκεί αυτό. Φυσικά αυτές οι διακήρυξεις είναι ένα σημαντικό μήνυμα που στέλνουμε στους ηγέτες ΑΣΕΜ, όμως ο ρόλος μας ως ε, βουλευτές θα πρέπει να είναι πιο φιλόδοξος. Εκπροσωπούμε πολλά εκατομμύρια πολίτες στην Ευρώπη και στην Ασία, πάρα πολλά εκατομμύρια θα έλεγα, και είμαστε η φωνή τους και περιμένουν από εμά να είμαστε πιο φιλόδοξοι στο να διαμορφώσουμε το μέλλον και να αντιμετωπίσουμε τις κοινέ προκλήσεις και στην Ασία, στην Ευρώπη, αλλά και σε όλο τον κόσμο εμεί, τα μέλη του Κοινοβουλίου, θα πρέπει να θετήσουμε την απαραίτητη νομοθεσία για να αντιμετωπίσουμε τι προκλήσει, να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και να προωθήσουμε την αηφόρο ανάπτυξη σε όλε τι διαστάσει, όπω το συζητάμε σήμερα καθώς ε, βλέπουμε να αυξάνεται η συνεργασία μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, υποστηρίζουμε και τις δικές σας προσπάθειες στην περιφερειακή ανάπτυξη και ενθαρρύνουμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να ακολουθήσουν την οδό της ε, συνεργασίας και της διπλωματίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πάντοτε υποστήριξε ισχυρά την ΑΣΕΜ και την ΑΣΕΠ και ενθαρρύνουμε τα ενδιαφερόμενα μέρη να ε, ενδυναμώσουν τις σχέσεις τους μεταξύ Ευρώπη και Ασία. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη συνδεσιμότητα μεταξύ των υπήρων μα, ε, να δημιουργήσουμε δεσμού μεταξύ των ανθρώπων, να αυξήσουμε τι ευκαιρίε για το εμπόριο, να δυναμώσουμε το διάλογο για την ασφαλεία και να συνεργαστούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά, η αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων τη κλιματική αλλαγή, χωρί χρονοτριβή, είναι ένα από τα επίγοντα θέματα για το μέλλον. Πρέπει να ε, φροντίσουμε να μεταμορφώσουμε τι οικονομίε μα, σε βιώσιμη βάση και να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ενεργειακής απόδοσης, της απόδοσης των πόρων, προκειμένου να έχουμε ένα υφόρο μέλλον για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Επομένως, θα ήθελα να ευχηθώ μια πολύ καρποφόρο συζήτηση. Θα διακηρύσω την έναρξη της 10ης κοινοβουλευτικής ε, συνάντησης της Εταιρικής Σχέσης Ασίας Ευρώπης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και για την προσοχή σας. Άρχεται η συνεδρίαση. Thank you for that very kind welcome and, and thank you for your... Ευχαριστούμε πολύ για το καλωσόρισμα. Ευχαριστώ και για την ε, Προεδρία σας στη Συντακτική Επιτροπή σήμερα το πρωί. Κάναμε πολλή δουλειά. Θα το ξαναδούμε το κείμενο βεβαίω και στην οριστική του μορφή αύριο. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ για πρώτη φορά στι Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και καθώ ε, ξεκινήσαμε πολύ καλά το πρωί, θα ξεκινήσουμε με το πρώτο θέμα που είναι η δήλωση του κυρίου Γιόντον Περενλέη Μπάνταρ Πελέικ, πρόεδρο του, της Επιτροπής Πολ, Δημόσιας Πολιτικής Εκπαίδευσης Πολιτισμού και Επιστημών ε, του Κοινοβουλίου της Μογγολίας, της χώρας που φιλοξένησε την τελευταία ΑΣΕΠ. Κύριε Μπατάρ Μπιλέκ, έχετε το λόγο. Αξιότιμε πρόεδρε Ταγιάννη, αξιότιμα μέλη των κοινοβουλίων της Ευρώπης και της Ασίας. Είναι μεγάλη μου χαρά που εκπροσωπώ την Μογγολία και συμμετέχω σε αυτή τη δέκατη συνάντηση κοινοβουλευτικής εταιρικής σχέσης Ευρώπης Ασία μαζί με όλου εσά τους ηγέτε από την Ευρώπη και την Ασία. Το ζήτημα της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής θεωρείται ένα από τα μείζωνα θέματα που απασχολούν τον κόσμο ολόκληρο τον τελευταίο, τα τελευταία χρόνια και απαιτεί συνεργασία. Σήμερα η Ευρωασιατική Διάσκεψη αποτελεί μια πολύ σημαντική πλατφόρμα που είναι ζωτική σημασία όχι μόνο για τη συνεργασία μεταξύ των δύο υπήρων αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο. Η Κοινοβουλευτική Διάσκεψη Ευρώπης-Ασίας αποτελεί σημαντικό στοιχείο της εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο ε, υπήρων και βοηθά στην επίτευξη συνένεσης σε μια σειρά αποζητήματα μεταξύ των δύο Υπήρων. Η Μογγολία προσπαθεί να συμμετέχει ενεργά σε αυτήν την εταιρική σχέση και στον διάλογο που διεξάγεται στο πλαίσιο αυτής. Όπως γνωρίζετε, η Μογγολία φιλοξένησε την, με επιτυχία την ε, ένατη ΑΣΕΠ και την ε, συνάντηση κορυφής με τίτλο εταιρική σχέση μέσω της ε, συνδεσιμότητας. Θεωρούμε ότι είναι σημαντική η 20η επέτειος από τη διακήρυξη της ε, Ουλάν Μπατόρ και πολύ σημαντικό το έργο που μας περιμένει στην τρίτη δεκαετία. Σημαίνει Θέλουμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο στον, ε, στις πολυπολικές σχέσεις και στην πολυμέρεια. Αυτή τη στιγμή έχουμε λοιπόν συναντηθεί εδώ για να συζητήσουμε πώς η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει την οικονομία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη μετανάστευση και την ασφάλεια σε ολόκληρο τον κόσμο. Και θέλουμε να δράσουμε ε, προς την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Αυτά τα ζητήματα απασχολούν και εμάς στη χώρα μου σήμερα. Ε, οι Μογγόλοι αντιμετωπίζουν ε, περίπλοκα προβλήματα και ζητήματα. Πρέπει να διδαχθούμε λοιπόν πώς θα ε, αξιοποιήσουμε τους φυσικούς πόρους, πώς θα, γίνουν, πώς θα επιτύχουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και βιώσιμες επενδύσεις. Το Κοινοβούλιο της Μογγολίας θέλει να διευρύνει και να ενισχύσει τις διακοινοβουλευτικές του σχέσεις με άλλα κοινοβούλια και πάντοτε συμμετέχει ενεργά και συμβάλλει σε αντίστοιχες ε, διαδικασίες σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Εμείς θέλουμε να προωθήσουμε και να αναπτύξουμε μια πιο ρεαλιστική συνεργασία η οποία θα αποφέρει αποτελεσματικότητα αποτελέσματα ρεαλιστικά όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των δύο υπήρων μας. Γι' αυτό και η Μογγολία ε, ε, αποδίδει μεγάλη σημασία στην ε, εταιρική σχέση την κοινοβουλευτική μεταξύ Ευρώπης Ασίας. Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της συνάντησής μας. Ευχαριστώ. Θέλω τώρα να καλέσω ε, την ε, κυρία Σιρίν Σάμιν, την ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου του Μπαγκλαντές, να λάβει το λόγο. Κύριε Συμπρόεδρε, κυρία Χαουτάλα, κύριε Ράιεν, Αντιπρόεδρε της Βουλής της Ρουμανίας, αντιπρόεδρε της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δούμας, πρόεδρε του Κοινοβουλίου της Φιλανδίας και του Βιετνάμ. Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να παρίσταμε στην 10η ε, Σύνοδο της Κοινοβουλευτικής Εταιρικής Συνεργασίας Ασίας Ευρώπης στις Βρυξέλλες. Η σύνοδος ε, αυτή, η εταιρική αυτή η σχέση προάγει τον απευθείας διάλογο μεταξύ κοινοβουλίων στην Ασία και την Ευρώπη. Χαίρομαι διότι εκπροσωπώ την Βουλή του Μπαγκλαντές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαστε μια χώρα η οποία πλήττεται σοβαρά από την μεταβολή του κλίματος. Είμαι βουνόμων στην ΑΣΕΠ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργανώνουν τη σημερινή μας σύνοδο. Σήμερα θα εστιαστούμε στην μεταβολή του κλίματος και τις συναφείς προκλήσεις τις επιπτώσεις ε, δηλαδή σε τρεις διαφορετικούς τομείς, την ασφάλεια, την μετανάστευση και την οικονομία. Αυτά θα συζητήσουμε σήμερα. Η μεταβολή του κλίματος αποτελεί σοβαρότατη απειλή κατά του πλανήτη. Επηρεάζει τις ζωές μας με τρόπο πολυσύνθετο και έχει και άλλες επιπτώσεις στην οικονομία. Η μεταβολή του κλίματος αφορά την ατμόσφαιρα, το έδαφος, τα τρόφιμα, την στέγη για δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πρέπει λοιπόν να διασφαλίσουμε μέτρα για την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι καιρός τα κοινοβούλια της Ασίας και της Ευρώπης να συνεργαστούν και να συμπήξουν μια εταιρική σχέση για να προαγάγουν περαιτέρω περιφερειακά σχέδια και στρατηγικές μέσω της αποτελεσματικής παγκόσμιας συνεργασίας. Πρέπει να αναγνωρίσουμε και να τονίσουμε ότι ο πολυμερής διάλογος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε από κοινού τι κοινέ μεγάλε προκλήσει, τη φτώχεια, τη μεταβολή του κλίματο, την ασφάλεια εφοδιασμού σε τρόφιμα, την επίλυση διαφορών, τα θέματα μετανάστευση, το προσφυγικό, πέραν των εθνικών συνόρων. Σε έναν όλο και περισσότερο αλληλοσυνδεδεμένο κόσμο, η συνεργασία είναι εκ των Ανουκάνευ Η ιατρική σχέση, η κοινοβουλευτική ιατρική σχέση Ασία Ευρώπη φέρνει κοντά τα κοινοβουλιά μας και εμείς ως ε, βουλευτές και εκπρόσωποι των λαών έχουμε λάβει την αποστολή να κάνουμε θετικές αλλαγές για τους λαούς που εκπροσωπούμε. Ο έλεγχος επί της εκτελεστικής εξουσίας μας δίνει τη δυνατότητα να, να φτιάξουμε ένα κόσμο ίσων ευκαιριών όπου καθένας μπορεί να πραγματοποιήσει τα όνειρά του έχουμε την δύναμη να αντιμετωπίσουμε και τη μεταβολή του κλίματο και τις επιπτώσεις της, να παράσουμε ασφάλεια στην καθημερινή ζωή για τους λαούς μας, να προστατεύσουμε το δικαίωμα στη ζωή με αξιοπρέπεια. Έχουμε ένα μοναδικό λοιπόν ρόλο. Μπορούμε να επηρεάσουμε θετικά τη ζωή των ανθρώπων στην Ασία και στην Ευρώπη για σήμερα και το μέλλον. Ας ενωθούμε και συλλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας στην πράξη για έναν καλύτερο πλανήτη για όλους. Πρέπει να θεσπίσουμε πολιτικές και να νομοθετήσουμε ως κοινοβούλια για να διασφαλίσουμε ότι θα πορευτούμε μαζί ως μια μεγάλη παγκόσμια οικογένεια χωρίς αποκλεισμούς. Ας ενώσουμε τις προσπάθειές μας να αυξήσουμε τη δυνατότητά μα να αντιπεξέλθουμε στη μεταβολή του κλίματο, να μειώσουμε τι εκπομπέ αερίων του θερμοκηπίου, να κάνουμε την οικονομία μα πιο πράσινη και πιο ανθεκτική. Η κοινοβουλευτική εταιρική συνεργασία Ασία και Ευρώπη θα προάγει επίση την κοινοβουλευτική διπλωματία. Νομίζω πετύχαμε διάφορα. Έχουμε ένα πλαίσιο ήδη στο Παρίσι, το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί και στην πράξη. Πρέπει επίση να πείσουμε όλους τους εμπλεκομένους να λάβουν μέτρα για να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη. Ας ψώσουμε λοιπόν την φωνή μας στο πλαίσιο των δεσμεύσεων των Παρισίων για να πετύχουμε και τους στόχους της εφορικής ανάπτυξης του 2020 για το καλό και της παγκοσμίας οικονομίας. Το Μάγκλαντες πιστεύει ότι η υλοποίηση στην πράξη της Συμφωνίας των Παρισίων είναι κοινή ευθύνη για την ευημερία του πλανήτη. Αυτό είναι το κλειδί. Χρειαζόμαστε όμω και χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου για το κλίμα, το οποίο δεν διαθέτει επαρκή χρηματοδότηση σήμερα. Οι στόχοι λοιπόν δεν θα επιτευχθούν χωρίς επαρκή και διαφανή χρηματοδότηση. Οι σχέσεις εμπιστοσύνη είναι πολύ σημαντικέ επίση. Πέρασαν ήδη τρία χρόνια το Παρίσι και ακόμη αισθανόμαστε την ανάγκη να επιταχύνουμε τον την ταχύτητα της υλοποίηση. Χρειάζεται επίση υποστήριξη των πλέον ευάλωτων χωρών σε χρηματοδότηση, τεχνολογία, τεχνογνωσία. Είναι σημαντικό για τις λιγότερο αναπτυγμένες χώρες και τις πιο ευάλωτες χώρες, κατά κύριο λόγο, να επωφεληθούν από τους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς των Παρισίων. Χρειαζόμαστε και άλλους τέτοιους μηχανισμούς με απλούστευμένες διαδικασίες. η Συμφωνία των Παρισίων πρέπει να γίνει λειτουργική και εφαρμόσιμη στην πράξη. Πιστεύω ότι η Συνοδός μας, η ΑΣΕΠ, μέσω της αμοιβαίας επικοινωνίας και μάθησης θα συμβάλλει στο να κάνουμε εν τέλει τη διαφορά. Η γη δεν είναι απλώς ένας πλανήτης, η γίνεται το σπίτι μας. Ας ενώσουμε τις προσπάθειές μας όλοι ανά τον πλανήτη για να κάνουμε αυτό το σπίτι μας πιο ασφαλές. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ, Dr. Σόντρι. Πολύ καλά προχωράμε. Θα έχουμε και τελική δήλωση και θα μπορέσουμε να έχουμε και πρόσθετες ε, δηλώσεις ε, από το βήμα. Αυτό το λέω για όσους θέλουν να κάνουν μια πρόσθετη δήλωση πριν ε, να ολοκληρώσουμε στις 11.30. Τώρα θα καλέσω... Ε, τον ε, αντιπρόεδρο της ε, Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων από την Κίνα να απευθυνθεί στην Επιτροπή μας. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, εκ μέρους του Κογκρέσου, του Εθνικού Κογκρέσου των Λεών της Κίνας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη οργάνωση αυτής της σημαντικής συνεδρίασης καθώς ε, και την ευγνωμοσύνη μας ε, για την ταχύτατη προετοιμασία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η δέκατη συνάντηση ΑΣΕΠ είναι το πρώτο παράπλευρο γεγονός και αποτέλεσμα της 12ης ε, διάσκεψης ΑΣΕΜ καθώς ε, όλος ο κόσμος αντιμετωπίζει σημαντικές αλλαγές, ε, περιβαλλοντικά θέματα και παγκόσμια κλιματική αλλαγή έχουν ε, πολύ μεγάλο αντίκτυπο στους ανθρώπους και την επιβίωσή τους. Η κλιματική αλλαγή και οι φυσικές καταστροφές έχουν επίπτωση ε, όχι μόνο στο φυσικό περιβάλλον, από το οποίο όλοι εξαρτώμαστε για την επιβίωσή μας, αλλά έχουν οδηγήσει και σε μία σειρά προβλημάτων, όπως ακραία καιρικά φαινόμενα, μείωση της ε, παραγωγής των τροφίμων, ε, έλλειψη νερού και ακόμη και πιο σοβαρές συνέπειες όπως και ο εκτοπισμός ανθρώπων και ξηράξεις. Πέρσι το καλοκαίρι όλο το βόρειο ημισφαίριο από μέχρι τον αρκτικό κύκλο ε, καλύφθηκε από κύματα καύσωνα σε πάρα πολλέ περιοχέ είχαμε υψηλέ θερμοκρασίε ρεκόρ. Ακραία καιρικά φαινόμενα όπω η ξηρασία, ε, κάποιες ε, ξαφνικές πυρκαγιές και ε, καταστροφικές καταιγίδε σάρωσαν την ασιατική ήπειρο. Αυτό μας έδειξε ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι πρόβλημα για τις μελλοντικές γενναίες, αλλά μια απειλή που όλοι αντιμετωπίζουμε σήμερα. Επομένως, χωρίς χρονοτριβή πρέπει να αναλάβουμε δράση για να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά θέματα. Γι' αυτό θέλω να αναφέρω τις εξής προτάσεις. Καταρχήν, θα πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις προσπαθίες μας για να ε, οικοδομήσουμε ένα κοινό μέλλον για την ανθρωπότητα. Αυτός ο πλανήτης είναι το μόνο σπίτι για την ανθρωπότητα. Όλες ε, οι χώρες ε, είναι στην ίδια κατάσταση ως μια κοινότητα με κοινό μέλλον. Αν έχουμε παροχημένες αντιλήψεις ε, όπως ο λιτερισμός και ε, ουσιαστικά δεν ε, αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας, θέλουμε περισσότερο με λιγότερη ευθύνη, τελικά θα βλάψουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Ε, θα πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Μόνο ε, αν συνεργαστούμε για να οικοδομήσουμε ένα παγκόσμιο σύστημα διακυβέρνησης που να είναι δίκαιο και ισότιμο και να βασίζεται σε συνεργασία μπορούμε να προσφέρουμε έναν ωραίο κόσμο για τις μελλοντικέ γενιές. Δεύτερον, θα πρέπει να λειοποιούμε τις ε, κοινέ μας υποχρεώσεις και να τηρούμε τους διεθνείς ε, κανόνες. Η Συμφωνία των Παρισίων ε, είναι μια συμφωνία ορόσημο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Δεν θα πρέπει να εγκαταλειφθεί καθώς ήταν δύσκολο να επιτευχθεί έχουμε διάφορες ε, κατανεμημένες ευθύνες και πρέπει να αναλάβουμε ε, τις ευθύνες αυτές ε, για να πετύχουμε τους διαφοροποιημένους στόχους. Και Φυσικά και η περιοχή της Ευρώπης και της Ασίας ε, θα πρέπει να υλοποιήσουν τη δεσμεύση τους ε, παρέχοντας οικοδόμηση ικανοτήτων ενώ από τις όμενες χώρες ε, θα πρέπει να βοηθήσουν η μία την άλλη και ενεργά να προωθήσουν τη συνεργασία νότου-νότου στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τρίτον, θα πρέπει να προβούμε, να επιδιώξουμε κοινές, κοινή ανάπτυξη και ε, περαιτέρω συνέργειες για την κοινή ανάπτυξη. Το, καθώς ε, μια μεγάλη τάση είναι η πράσινη οικονομία, κλιματικές ε, δράσεις και οικονομική ανάπτυξη αμοιβαία αλληλοενισχύονται θα πρέπει να δούμε το θέμα της πράσινης χρηματοδότησης και Τη εμπορία του άνθρακα. Αυτά παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στο να προωθήσουν την οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει να συντονίσουμε την αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και την εφαρμογή της ε, ατζέντα ε, για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030. Δεν ε, θα πρέπει να έχουμε οικονομική ανάπτυξη βάρος του περιβάλλοντος και να αγνοήσουμε ε, την, ε, τα δικαιώματα του ανθρώπου για επιβίωση. Δεν είναι σοφό κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να έχουμε μια κοινή ασφάλεια κατά των κινδύνων που θέτουν η κλιματική αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Θα πρέπει να έχουμε ένα νέο όραμα για την ασφάλεια. Ένα όραμα το οποίο ε, θα περιλαμβάνει ε, μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ασφάλεια. Χρειαζόμαστε ολιστικά και συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να προωθήσουμε ρεαλιστική συνεργασία και να δομήσουμε προβλήματα της διατροφικής ασφάλειας, ανθρωπιστικής κρίσης και μαζικών προσφυγικών ροών αλλά και άλλων κινδύνων ασφαλείας που μπορεί να προκύψουν από την κλιματική αλλαγή. Οι αναπτυγμένες χώρες και οι σχετικοί διεθνεί οργανισμοί θα πρέπει να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους, να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες, να ενδυναμώσουν την ικανότητά τους στο να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγέ, να χαράξουν στρατηγικές μετριασμού ε, των κλιματικών αλλαγών, ε, να ε, μπορέσουν να μειώσουν τους κινδύνους, να βελτιώσουν την διαχείριση του μεταναστευτικού και να χτίσουν ανθεκτικότητα. Ως αναπτυσσόμενη χώρα έχουμε πάνω από ένα ε, δισεκατομμύριο, 300 εκατομμύρια ανθρώπους και είμαστε αυτοί που υποφέρουμε περισσότερο από τον αντίκτυπο της κλιματικής ε, αλλαγής η Κίνα, ε, καταπολεμώντας την κλιματική αλλαγή, δεν κινείται μόνο βάσει της απέτησης για βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και βάσει τη δέσμευσή μα να παίξουμε και το δικό μας ρόλο στην παγκόσμια κλιματική διακυβέρνηση. Η Κίνα έχει πάρει διάφορα μέτρα όπως ε, παραδείγματος χάρη την αναβάθμιση των εθνικών ε, υποδομών και του ενεργειακού μείγματος. Ε, αναπτύσσει πράσινη αρχιτεκτονική και μεταφορές χαμηλού άνθρακα δημιουργεί μία αγορά ανταλλαγής δικαιωμάτων εκπομπών και προωθεί την πράσινη οικονομία το Κογκρέσο δίνει πολύ, σημαντική, πολύ μεγάλη σημασία στην κλιματική αλλαγή και υιοθετεί νόμους όπως ε, έχει να κάνει ε, με την νομοθεσία για την ε, εξοικονόμηση ενέργειας, το νόμο για τα δάση, το νόμο για την ατμοσφαιρική ρήπανση κτλ. Επίσης εργαζόμαστε για επί ενός νομοσχεδίου για την κλιματική αλλαγή. Χάρη στις προσπάθειές μας έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Τα τελευταία πέντε χρόνια η κατανάλωση ενέργειας και νερού μονάδα ΑΕΠ στην Κίνα έχει μειωθεί πάνω από 20% η αναλογία της ε, συνκατανάλωσης έχει μειωθεί κατά 1,8%. Το μερίδιο της κατανάλωσης καθαρής ενέργειας έχει αυξηθεί κατά 6,3%. Η κάλυψη των δασών έχει αυξηθεί κατά 10,87 δισεκατομμύρια εκτάρια και ο αριθμό των ημερών ε, όπου έχουμε πολύ μεγάλη ατμοσφαιρική ρήπανση στις πόλεις έχει μειωθεί κατά 15%. Η πράσινη ανάπτυξη δίνει στην Κίνα μια πολλά υποσχόμενη προοπτική. Η Κίνα παίζει ένα σημαντικό ρόλο ε, στο ε, να ε, θα σπίσει διεθνή συνεργασία κατά της κλιματικής αλλαγής. Έχει γίνει ηγέτης ε, στην ε, οικολογική ανάπτυξη. Έχει συμμετέχει ενεργά η κινέζικη κυβέρνηση στο να διευκολύνει την Συμφωνία των Περισσίων και την έχει υπογράψει. Εμείς τιμούμε τις δεσμεύσεις μας και θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τη συμφωνία με πολύ μεγάλη προθυμία κάνοντας ορθή χρήση ε, της ε, πλατφόρμας όπως ε, είναι η πρωτοβουλία «Μία ζώνη, μία οδός» και ενισχύοντας τη συνεργασία νότου-νότου ενισχύουμε τη συνεργασία μας με όλες τις χώρες για την κλιματική αλλαγή στην οδό της βιώσιμης ανάπτυξης. Το 2013 ο πρόεδρος Σι ανακοίνωσε ότι η διάσκεψη της κλιματικής αλλαγής ε, στο Περισσίον, η Κίνα, θα ε, δημιουργούσε σχέδια συνεργασίας ε, για να δημιουργήσει 10 βιομηχανικά πάρκα με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και να ξεκινήσει άλλα προγράμματα προσαρμογής σε άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, δίνοντας διάφορες ευκαιρίες κατάρτισης για την κλιματική αλλαγή. Εμείς ε, για πλαίσια αυτών των προγραμμάτων έχουμε υπογράψει μνημόνια συνεννόησης και παρέχουμε ε, μέσα καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής ε, στο Βιετνάμ, στις Φιλιππίνες, στη Μιανμάρ, στη Μογγολία και σε άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι, οι χώρες της Ευρασίας είναι θύματα της κλιματικής αλλαγής αλλά και συμμετέχοντες στις δράσεις για το κλίμα. Ε, στην επόμενη 12η διάσκεψη ΕΣΕΜ αναμένουμε οι ηγέτες ε, να ε, μπορέσουν να επαναλάβουν τις δεσμεύσεις τους για την επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και να υπάρξει μεγαλύτερη συνεργασία στην ανάληψη στόχων για το κλίμα. Η Κίνα είναι έτοιμη να ενώσει τις προσπάθειές της με τις ε, χώρες της Ευρασίας για να ανταλλάξουμε εμπειρίες που σχετίζονται με την περιβαλλοντική διακυβέρνηση και την οικονομική ανάπτυξη, να διατηρήσουμε μια ενεργή συμμετοχή στην πολυμερή διακυβέρνηση της κλιματικής αλλαγής, έτσι ώστε από κοινού να μπορούμε να οικοδομήσουμε μια, έναν ανοιχτό συμμετοχικό κόσμο όπου θα έχουμε διαρκή ειρήνη, παγκόσμια ασφάλεια και ευημερία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τσάνγκ. Έχουμε λίγα λεπτά προτού περάσουμε στην πρώτη θεματική συζήτηση. Αν κάποιος θέλει το λόγο για να τοποθετηθεί, μπορεί να το κάνει τώρα. Ε, προτού ξεκινήσουμε με την ε, θεματική συνάντησή μας. Δεν βλέπω κάποιον να ζητά το λόγο. Οπότε θα δώσω το λόγο στην κυρία Χάουταλα για να ξεκινήσει η θεματική συζήτηση, η πρώτη και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ράιαν και τώρα έχω τη χαρά να ξεκινήσουμε την συζήτηση για την κλιματική αλλαγή, την πρόκληση για τις πολυμερείς σχέσεις. Χαίρομαι πάρα πολύ που ακούσαμε ήδη τόσες πολύτιμες παρεμβάσεις στη συζήτηση αυτή. Έχω τη χαρά λοιπόν τώρα να καλέσω τους ομιλητές μας να ανέβουν εδώ στο βήμα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώ Λάινεν που είναι ο εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κλιματική αλλαγή και είναι επίσης επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Κίνα. Είναι πραγματικά ο καταλληλότερος άνθρωπός μας για αυτή τη δουλειά. Έχουμε μαζί μας επίσης τον κύριο Σκοτ Ράιαν, πρόεδρο της Αυστραλιανής Γερουσίας. Μαζί μας έχουμε επίσης την κυρία Κάρμεν Ιλεάνα Μιχαλέσκου που είναι αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ε, του Ρουμανικού Κοινοβουλίου. Έχουμε μαζί μας τη Ρόζα Μαρία Ρομέρο Σάντζες... που είναι ε, αντιπρόεδρος της Γερουσίας της Ισπανίας και έχουμε μαζί μας και τον πρώτο αντιπρόεδρο ε, του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, τον κύριο Πεκαρίνεν. Θα ήθελα επίση να καλέσω στο βήμα τον κύριο Φουν Χοκιέν, αντιπρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης του Βιετνάμ και εκπρόσωπο του Ινδικού Κοινοβουλίου. Μόλις ανέβουν λοιπόν οι ομιλητές στο βήμα, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Να προτείνω μετά από αυτήν τη συζήτηση να βγάλουμε την οικογενειακή μας φωτογραφία σας παρακαλώ. Γι' αυτό ε, μη φύγετε από την αίθουσα μετά τη συζήτηση. So I'd like to um, Uh, ask that the speakers would uh, um, speak for about five... Λοιπόν, θα ήθελα να ζητήσω από τους ομιλητές να μην ξεπεράσουν τα 5 με 7 λεπτά, γιατί έχουμε αρκετούς. Θα υπάρχει αρκετός χρόνος το απόγευμα για να κάνουμε ανοιχτή συζήτηση στις, ε, στα θεματικά πάνελ που ε, διοργανώνουμε. Ο λόγος ε, στον κύριο Λάινεν, τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι από την Ασία και την Ευρώπη. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σήμερα την κλιματική αλλαγή ως ε, βασικό θέμα αυτής της ε, συνδιάσκεψης ΑΣΕΜ. Εγώ συμμετείχα στην COP1 το 1995 στο Βερολίνο μετά την ε, διάσκεψη του Ρίου του Τζανέιρο και τώρα πλέον βρισκόμαστε εν ώψη της COP 24 στο Κατοβίτσε. Πέρασαν πολλά χρόνια και ευτυχώς υπάρχει πλέον παγκόσμια συνένεση, λίγος πολύ, ότι το πρόβλημα της αντιμετώπισης της, ε, υπερθέρμανσης του πλανήτη είναι κοινός στόχος που αφορά όλα τα έθνη του κόσμου. Δυστυχώς σε αυτή τη φάση που ε, χρειαζόμαστε πιο πολύ από ποτέ τις πολυμερείς σχέσεις υπάρχουν κάποιοι που επιτίθενται στην πολυμέρεια και θέλουν να ακολουθήσουν έναν απομονωμένο δρόμο. Και αυτό είναι πραγματικά δυστύχημα γιατί το κλίμα, η ατμόσφαιρα είναι κοινό μας αγαθό όλων των λαών, ανήκει στην ανθρωπότητα είναι ένα παγκόσμιο αγαθό που ανήκει σε όλους μας. Δεν ανήκει σε κανέναν ξεχωριστά. Γι' αυτό χαίρομαι που παρά το γεγονός ότι η Αμερικανική κυβέρνηση εξήλθε τη Συμφωνία των Παρισίων, όλες οι άλλες κυβερνήσεις του κόσμου έχουν επιβεβαιώσει ότι συνεχίζουν την εφαρμογή της συμφωνίας αυτής. Θεωρώ ότι η Ευρώπη και η Ασία για διαφορετικούς λόγους έχουν ε, πολύ μεγάλες ευθύνες. Η Ευρώπη, διότι συνέβη πριν από 200 χρόνια εδώ να ξεκινήσει η εκβιομηχάνηση, η οποία... Ε, μεταφέρθηκε και σε ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο μαζί με το οικονομικό μοντέλο που γέννησε και ξέρουμε ότι πλέον αυτό το οικονομικό μοντέλο πρέπει να αλλάξει. Σε λίγα χρόνια ο πληθυσμός της γης θα αγγίξει τα 10 δισεκατομμύρια και αυτό φυσικά πρέπει να επηρεάσει και το οικονομικό μοντέλο που ε, εφαρμόζουμε. Στην Ασία επειδή ε, υπάρχουν αναπτυσσόμενες οικονομίες και ο μεγαλύτερος πληθυσμός του πλανήτη είναι αναγκαίο να περάσουμε σε μέτρα εξυγχρονισμού και αναβάθμισης. Μια δουλειά που όμως έχει ξεκινήσει και που είναι πολύ ελπιδοφόρα. Ε, Ξέρετε ότι και εμείς έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες μας όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έχουμε ήδη οδηγίες για τα κτίρια, την ενεργειακή αποδοτικότητα, τις, τις μεταφορές. Τώρα βρισκόμαστε στη φάση αντιμετώπισης ε, των ε, εκπομπών από τα αυτοκίνητα για να καταλήξουμε σε αυτοκίνητα, σε οχήματα χαμηλών εκπομπών. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλο μέρος της δουλειάς που μας αναλογεί για την επόμενη δεκαετία και γι' αυτό ο Επίτροπος ε, υπεύθυνο για το κλίμα ήταν σε θέση να ε, ανακοινώσει ότι θέλουμε μάλιστα να ενισχύσουμε τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει στο Παρίσι και να επιδιώξουμε ακόμα υψηλότερους στόχους. Εμείς ε, έχουμε δεσμευτεί να μειώσουμε κατά 40% το διοξίδιο του άνθρακα ε, έως το 2030 ε, και πλέον ετοιμάζεται νομοθεσία η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα να μειώσουμε κατά 45% τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Έχοντας υπόψη ότι θα υπάρξουν και φάσεις ε, και αποφάσεις αναθεώρησης το 2023. Υπάρχει λοιπόν ακόμη αρκετός χώρος και χρόνος για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας. Ε, εγώ ήμουν εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ε, κλιματική διπλωματία. Και όταν κανείς μιλά για πολυμερείς σχέσεις, προφανώς και χρειάζονται και διπλωματικές συμφωνίες. Δεν μπορεί κανείς να αναγκάσει κάποιον άλλον να κάνει κάτι, πρέπει να πείθει κανείς. Ε, και στη συνέχεια να ελπίζει ότι όλοι θα ακολουθήσουν το ασυμπεφωνηθέντα. Η κλιματική δράση σε ενωσιακό επίπεδο λοιπόν, σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει ότι θέλουμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας σε ολόκληρο τον κόσμο των αντιπροσωπιών της ευρωπαϊκή ένωση για να βρούμε εταίρους για καθαρή ενέργεια, για καθαρές τεχνολογίες, για ε, αντίστοιχες συμμαχίες, για καινοτόμες και ε, πρωτοπόρες ομάδες σε κυβερνητικό επίπεδο, σε εταιρικό επίπεδο, σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών. Εμείς λοιπόν έχουμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να εξορθολογήσουν και να εντάξουν, να συμπεριλάβουν την κλιματική πολιτική σε όλες τις άλλες πολιτικές μας. Τη βιομηχανική πολιτική, την εμπορική πολιτική που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, πολιτική για την ανάπτυξη, για τη γεωργία και Νομίζω λοιπόν ότι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά βρισκόμαστε στη φάση έναρξης μιας νέας περίοδου ενίσχυσης των προσπαθειών μας. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας, χαίρομαι, την την... χαίρομαι πολύ για την παρουσία σας εδώ και πιστεύω πραγματικά ότι η Ευρώπη και η Ασία είναι οι δύο πυλώνες που θα οδηγήσουν και θα καθοδηγήσουν την πρόοδο του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ ε, λοιπόν για όλα όσα κάνετε γιατί είναι πολύ σημαντικά ε, όλα αυτά που θα κάνουμε σήμερα για τις ε, επόμενες γενιές, τις γενιές του μέλλοντος. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. πολύ ενδιαφέρον που ήσουν στην COP1. Ήμουν στην COP2 στο Κιώτον, δεν κάνω λάθος. Και τώρα, ο συμπροεδρός μου συνεχίζει εκ μέρους της ε, γερουσίας της Αυστραλίας, ε, Σκοτ. Και Σκοτ Ράιαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, εισαγωγή. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά όλους και έχω θα έχω την τιμή να πω λίγα λόγια για τη μεταβολή του κλίματος η οποία συνεπάγεται οικονομικούς κινδύνους που θα ενταθούν την επόμενη δεκαετία. Θα είναι μια πολυμερής πρόκληση. Τον Μάιο η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνα στην Γερουσία μα εξέδωσε έκθεση για τι επιπτώσει τη μεταβολή του κλίματο στην Αυστραλία. Η έκθεση διαλαμβάνεται των κινδύνων αλλά και των ευκαιριών. Διαπιστώσαμε ότι διατρέχουμε και κινδύνους ασφαλείας. Διότι η μεταβολή του κλίματος οξύνει τις προκλήσεις για το περιβάλλον, τα ύδατα, τα τρόφιμα και την υγεία. Το περιβάλλον μεταβάλλεται, όπως είπαν και οι προηγούμενοι μιλητές, και αυτό σημαίνει ότι οξύνονται και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτές οι προκλήσεις σημαίνουν λιγότερη σταθερότητα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν και σε σειράξεις ή κύματα μετανάστευσης. Πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στο φαινόμενο, να συζητήσουμε τα θέματα ασφάλεια, Πολύ μάλλον καθώς κάποιες κοινότητε θα γίνουν ακόμα περισσότερο ευάλωτε, ιδιαίτερα σε νησιά. Αυτέ απειλούνται περισσότερο, απειλείται η καθημερινή του ζωή και επιβίωση. Η πολιτική σταθερότητα στον ειρηνικό προποθέτει οικονομική σταθερότητα. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει η Αυστραλία να προστατεύσει τα δικά τη οικονομικά συμφέροντα αλλά και αυτά τη περιοχή. Διάφορε αυτές οι κυβερνήσεις έχουν αναγνωρίσει ευκαιρίες και κινδύνους. Μια πρόσφατη λευκή βίβλος του Υπουργείου Εξωτερικών της Αυστραλίας εστιάζει στις απειλές κατά της εφορικής εξασφάλισης τροφίμων και άλλων πόρων. Υπάρχουν λοιπόν απειλές οι οποίες ε, προποθετούν συντονισμό σε πολυμερές επίπεδο από τις χώρες μάχης για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, μια συντονισμένη πολυμερή απόκριση. Η Αυστραλία θα τηρήσει την Συμφωνία των Παρισίων μέχρι το 2030 θα μειώσει κατά 28% τις εκπομπές της και αυτό είναι λογικό, είναι εύλογο και συνάδει με αυτά που θα κάνουν και άλλες χώρες. Θα ενισχύσουμε λοιπόν την διεθνή δράση για το κλίμα, θα συμμετάσχουμε σε φόρα και συμφωνίες όπως η πλατφόρμα για τους εκτοπισμένους λόγω φυσικών καταστροφών και θα προσπαθήσουμε να μετριάσουμε τους ε, κινδύνους μέχρι το 2030. Η απόκρισή μας σημαίνει ότι θα εντείνουμε και την αναπτυξιακή βοήθεια. Ένα δισεκατομμύριο θα πληρώσουμε σε περίοδο 5 ετών σε αναπτυσσόμενες χώρες με γνώμονα τους κινδύνους από την μεταβολή του κλίματος. Το φαινόμενο εντείνει πολλαπλούς κινδύνους. Το προϋποθέτει λοιπόν νέα διακυβέρνηση για τα δάση, για τα ύδατα, για τις υποδομές και περισσότερες πολυμερείς προσπάθειες. Θα ήθελα να κλείσω τονίζοντας ότι η Ασία διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στα θέματα αυτά. Εμείς ως βουλευτές, ως κοινοβούλια διαδραματίζουμε μεγάλο ρόλο στην εξασφάλιση συνένεση στην απόκριση και στην θέσπιση προτεραιοτήτων. Διότι πολλά από αυτά τα θέματα θα πετήσουν μακρόχρονη, μακροπρόθεσμη δράση. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε για μια φορά την ευκαιρία να μιλήσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ράιαν. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στην κυρία Κάρμεν Λεάννα Φαλσέσκου, η οποία είναι αντιπρόεδρος ε, της Βουλής της Ρουμανίας. Να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μου δίνετε να κάνω μια παρουσίαση. Όλοι γνωρίζουμε ότι η κλιματική αλλαγή είναι παγκόσμια πρόκληση με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ασφάλεια των χωρών. Πρόκειται για μια απειλή κατά της παγκόσμιας σταθερότητας και ασφάλειας επειδή έχει ε, συνέπειες και στους ανθρώπους όπως ε, είναι οι σειράξεις, ε, οι ασθένειες, οι εκτοπισμένοι κτλ. Αυτοί που αντιμετωπίζουν τους χειρότερους κινδύνους είναι οι πιο φτωχοί περιοχή με τους λιγότερους πόρους και την μικρότερη ικανότητα να ε, αντιμετωπίσουν την κρίση. Η ασφάλεια η κλιματική λοιπόν είναι πολύ σημαντική ε, στον ε, αλληλοσυνδεδεμένο κόσμο μας. Η δική μας ασφάλεια έγκυται στην ασφάλεια των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Το να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή μπορεί να σώσει ζωές ε, παγκοσμίω, ενώ θα διασφαλίσει ένα πιο ασφαλές μέλος. Η πραγματική η αποτελεσματική διαχείριση κλιματικής αλλαγής απαιτεί το να συμμετέχουν η κοινωνία των πολιτών, τα κράτη, οι επιχειρήσει και να υπάρξει συντονισμό σε διάφορα επίπεδα όπως εξωτερική, οικονομική, πολιτική, περιβαλλοντική και οικονομική συνεργασία. Θα πρέπει να διατηρήσουμε λοιπόν την όθηση και να θετήσουμε όλα τα στοιχεία που χρειάζονται για να καταστήσουμε επιχειρησιακή τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή και να εφαρμόσουμε τις δεσμεύσεις μας. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Ρουμανία έχει ε, κυρώσει την Συμφωνία των Παρισίων την 1η Ιουνίου 2017 έτσι ε, αναλαμβάνει τις δεσμεύσεις της, υποστηρίζει την Γαλλική Πρωτοβουλία σε ό,τι αφορά το Σύμφωνο για το Περιβάλλον και είναι ε, μεταξύ ε, των υπογραφών του ε, συμφώνου επιθετήθηκε από τον ΟΗΕ. Έχουμε ε, Διάφορε νομοθετήματα για την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή που υιοθετήθηκαν από το Κοινοβούλιο της Ρουμανίας είχαν υιοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συνεισφορά για τη Συμφωνία των Πορυσίων συμπεριλαμβάνεται στην ε, συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωση και των κρατών μελών που προωθήθηκε ε, στην γραμματεία της UNFCCC στις 6 Μαρτίου 2015 η Ρουμανία ακολουθεί ε, ε, τις προτάσεις και δεσμεύεται για την εφαρμογή τους. Έτσι θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Αν μου επιτρέπετε, πέρα από τα κυρία στοιχεία, θα ήθελα να τονίσω και κάποιες πτυχές ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τη Συμφωνία των Παρισίων. Καταρχήν, ε, μακροπρόθεσμο όραμα της ε, απαραίτητης μετάβασης. Με συγχωρείτε προκειμένου να έχουμε μια καλή επικοινωνία και σε άλλες χώρες. Μπορείτε να μιλήσετε κάπως πιο αργά. Αυτή είναι μια πρόταση σε όλους σας. Έχουμε διερμηνία υψηλού επίπεδου, όμως ε, είναι υπερβολική ταχύτητα μερικές φορές. Έχουμε χρόνο. Λοιπόν, αναφέρομαι σε κάποιες πτυχές που έχουν να κάνουν με τη Συμφωνία των Παρισίων. Καταρχήν το μακροπρόθεσμο όραμα της απαραίτητης μετάβασης ε, ε, στο να έχουμε λιγότερες εκπομπές στο αερίο του θερμοκηπίου στο, στον 21ο αιώνα μέσω της πρόθεσης της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξάλληψης της φτώχειας. Δεύτερον, η θέσπιση μακροπρόθεσμων στόχων στη Συμφωνία των Παρισίων να περιοριστεί η αύξηση της ε, παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου και ταυτόχρονα η υποστήριξη των κρατών στη Συμφωνία των Παρισίων για να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας ε, μέχρι 1,5 βαθμό Κελσίου ε, σε ό,τι αφορά το μέσο όρο παγκοσμίω. Τρίτον, ε, μέσω της εμπλοκής των αναπτυγμένων χωρών να διασφαλίσουμε την ενεργοποίηση οικονομικών πόρων για τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, και να διευκολύνουμε τη μεταφορά τεχνολογίας και να αυξήσουμε την ικανότητά τους να προσαρμοστούν ε, στα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής αλλά και να εφαρμόσουν μέτρα για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατόπιν αναγνώριση από τα κράτη που ε, καταρτίζουν πολιτικές για την κλιματική αλλαγή για την ανάγκη να συνεργαστούν και αυξήσουν την κατανόηση, τη δράση τους και την υποστήριξη σε διάφορους τομείς όπως είναι συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, ε, την ε, πρόληψη ε, κρίσεων ε, στην περίπτωση που έχουμε καταστροφές από τις κλιματικές αλλαγές. Επίσης, να αναπτύξουμε έναν στόχο παγκόσμιας ποιότητας για την προσαρμογή, προκειμένου να αυξήσουμε τη δυνατότητα προσαρμογής, την ανθεκτικότητα και να μειώσουμε την ευπάθεια. Τα κράτη θα πρέπει να αναπτύξουν σχέδια προσαρμογής ε, που θα τα κοινοποιούν ε, εγκαίρως με εφαρμοστικά μέτρα. Έκτο, προώθηση μιας παγκόσμιας διαδικασίας αξιολόγησης της πρόοδου σε ό,τι αφορά ε, την επίτευξη των στόχων βάσει συστημάτων παρακολούθησης και αναφοράς που διασφαλίζουν διαφάνεια και λογοδοσία και τέλος προώθηση ενό ενός κύκλου αναθεώρησης δεσμεύσεων με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα προκειμένου να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της Συμφωνίας των Παρισίων και ε, οι ε, δεσμεύσεις να μην είναι κάτω από τα εφιστάμενα επίπεδα φιλοδοξίας, αγαπητοί συνάδελφοι. Η Ρουμανία θα αναλάβει την ε, Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρώτο εξάμεινο του 2019. Ο κύριος στόχος ε, θα είναι να ε, προωθήσει ε, όλους τους φακέλους που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, να συνεχίσει τις προετοιμασίες για την COP24 και την προετοιμασία για τα θέματα που θα συζητηθούν και να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή του Παγκόσμιου Προγράμματος για την εφαρμογή της Συμφωνίας των Περισσίων που υιοθετήθηκε από την COP24. Σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή. Thank you very much, uh, Ευχαριστούμε κυρία Μιχαλσέσκου. Και τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Μάουρι Πεκαρίνεν, το πρώτο αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, τον περασμένο Οκτώβριο Οκτώβριο έκθεση του ΟΗΕ μας υπενθύμησε ότι τα κράτη έχουν επιτύχει μόλις το 1 τρίτο των όσων πρέπει να επιτύχουν έως το 2030. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε συλλογικές προσπάθειες προκειμένου να αλλάξουμε την ε, πορεία. Και αυτό αφορά όλους τις ανεπτυγμένες και τις λιγότερα ανεπτυγμένες χώρες. Υπάρχουν πολύ σημαντικοί και σοβαροί λόγοι για την υπερθέρμανση του πλανήτη και η σύμβαση πλαίσιο του ΟΗΕ του 1992 προέβλεπε διαχωρισμό των χωρών σε ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες και προέβλεπε υποχρεώσεις μόνο για τις ε, ανεπτυγμένες βιομηχανικές χώρες. Ωστόσο, οι συνθήκες έχουν αλλάξει δραματικά. Για παράδειγμα, οι εκπομπές της Κίνας ανέρχονται στο 27% των παγκόσμιων εκπομπών, ενώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στο 10%. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες του 1992 είναι σήμερα κάποιες από τις ε, πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Σύμφωνα λοιπόν με διεθνείς φορείς, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα στις ανεπτυσσόμενες χώρες έχουν τριπλασιαστεί από το 1990. Και πρέπει επίσης ε, και εμείς οι Ευρωπαίοι να μην ξεχνάμε ότι οι εκπομπές κατά κεφαλή παραμένουν πολύ υψηλές στην Ευρώπη. Υψηλότερε κατά πολύ από ό,τι για παράδειγμα στην Ινδία. Με τις δράσεις της όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποδείξει ότι μπορεί κανείς να σπάσει το συσχετισμό μεταξύ εκπομπών και ανάπτυξης. Με άλλα λόγια, οι εκπομπές στην Ευρώπη έχουν μειωθεί ενώ η οικονομία αναπτύσσεται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει την, προσήλωση, την προσήλωσή της να συνεχίσει σε αυτή την πορεία και τις προσπάθειες για την επίτευξη του στόχου του 2030 για 30% μείωση των εκπομπών έως το 2030. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης και για εμάς αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο. Η Συμφωνία των Παρισίων του 2015 μας γεμίζει ελπίδες είναι μια νομικά δεσμευτική σύμβαση η οποία προβλέπει παγκόσμια μέτρα και συλλογικέ δράσεις από όλε τις χώρες. Σκοπός είναι να περιοριστεί η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας του κόσμου σε επίπεδα χαμηλότερα από 2 βαθμούς Κελσίου και προβλέπεται συλλογικές ενέργειες και μέτρα για να αποτραπεί ε, αύξηση θερμοκρασίας υψηλότερη από αυτό το όριο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση μια σειρά από περιβαλλοντικές συμφωνίες. Σκοπός είναι να καταλήξουμε σε συμφωνία το Δεκέμβριο του 2018 στην COP24 ε, στο Κατοβίτσε της Πολωνίας. Ένα από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν είναι αν αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να είναι εξίσου υποχρεωμένες να υποβάλουν εκθέσεις σχετικά με τις εκπομπές τους και την ε, επίτευξη των στόχων. Κάποιες αναπτυσσόμενες χώρες πιέζουν για να διατηρηθεί ο διαχωρισμός του 1992. Αυτό όμως αντιβαίνει στο πνεύμα της Συμφωνίας των Παρισίων όπου επετεύχθη συμβιβασμός όσον αφορά τον διαχωρισμό αυτών. Αν η συμφωνία περιλαμβάνει τους ίδιους κανόνες για όλους, θα ε, επιβεβαιωθεί αυτό το, το πνεύμα συμβιβασμού που επετέφθη στο Παρίσι. Αυτή τη στιγμή όλες οι χώρες είναι υποχρεωμένες να μειώσουν τις εκπομπές τους, να υποβάλουν σχετικές εκθέσεις όσον αφορά την πρόοδο ε, που έχουν σημειώσει στην επίτευξη του στόχου αυτού. Πριν από ένα χρόνο, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε θα αποσυρθούν από τη Συμφωνία του Παρισιού. Ο πρόεδρος μάλιστα περιέγραψε την συμφωνία ως έξυπνη κίνηση που εξήφαναν άλλες χώρες για να υποσκάψουν την δύναμη και την ισχύ ε, των ΗΠΑ και εξέφρασε αμφιβολίες για τον τρόπο με τον οποίο καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία. Η Ευρώπη και η Ασία έχουν μεγάλα περιθώρια διμερούς συνεργασίας αλλά και σε πολυμερείς σχέσεις για να ε, προάγουν τις ε, τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό θα δώσει ε, πολύπλευρες ευκαιρίες σε πολλές χώρες των υπήρων μας, καθώς πολλές από τις χώρες μας είναι δραστήρια μέλη πολλών βιομηχανικών φορέων και οργανισμών. Θέλω λοιπόν να συζητήσουμε περαιτέρω για το πώς θα μπορέσουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία μεταξύ ευρωπαϊκών και ασιατικών χωρών στα ε, πολυμερή φόρα και μπορούμε να καθορίσουμε και ποια ε, φόρα είναι τα πλέον κατάλληλα για την ενίσχυση της συνεργασίας μας. Επιπλέον μπορούμε να συζητήσουμε τα ζητήματα που σχετίζονται με την συνεργασία στον τομέα της ε, τεχνολογίας της ενέργειας. Εμείς, ε, η, χώρα μου, η Φιλανδία, έχει πολλές σχέσεις με ασιατικές χώρες και έχουμε εμπειρογνωμοσύνη σε, σε τομείς όπως είναι τα βιοκαύσιμα, η βιοενέργεια και η παραγωγή της και παρεμπιπτόντως να σας πω ότι στη Φιλανδία οι μεταφορές ε, σήμερα ε, συμπεριλαμβάνουν μια διάσταση 20% ανανεώσιμων ποιών ενέργειας. Και αυτό είναι υποχρέωση, δεν ήταν τυχαίο, ήταν υποχρέωση η οποία έχει κατοχυρωθεί στην νομοθεσία μας και έτσι έχουμε επιτύχει το 20%. Εκτός από τα βιοκαύσιμα λοιπόν και τη βιοενέργεια, έχουμε έξυπνα δίκτυα και πυρηνική ασφάλεια. Αυτά είναι τα δυνατά μας σημεία, αν θέλετε. Και παρά το γεγονός ότι ε, είμαστε χώρα κοντά στον αρκτικό κύκλο, μπορώ να σας πω ότι είμαστε πρωτοπόροι και στην ηλιακή ενέργεια και έχουμε ερευνητικές και επιστημονικές ομάδες οι οποίες μάλιστα ε, έχουν ε, να επιδείξουν σημαντικά αποτελέσματα στο έργο τους. Αν υπάρξει λοιπόν ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο υπήρων μας και εγώ αυτό θα ήθελα, νομίζω ότι μπορούμε να, να επιτύχουμε ακόμα σημαντικότερα αποτελέσματα. Ο τομέας της χρήσης γης και τα δάση επίσης θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να τονίσω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο μέρος των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα προέρχεται από τη χρήση ορυκτών πηγών ενέργειας στις μεταφορές, στην ενέργεια αλλά και ε, ο τομέας της χρήσης γης είναι πολύ σημαντικός. Εμείς έχουμε μεγάλη πυρογνωμοσύνη όσον αφορά τη διαχείριση των δασών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Κάθε χώρα στον κόσμο είναι υπεύθυνη για τη βιώσιμη αξιοποίηση των φυσικών της πόρος χωρίς να ε, πλήττονται και να βλάπτονται ε, άλλες χώρες. Εμείς δεν βρίσκουμε το λόγο να προστατεύσουμε και να διατηρήσουμε μόνο τα δικά μας ε, δάση και να εγκαταλείψουμε τα δάση του υπόλοιπου πλανήτη. Ευχαριστούμε πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πεκαρίνεν. Κρατούμε την έκκληση για περισσότερη συνεργασία σε πολυμερή πλαίσια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης, ιδιαίτερα σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Πριν καλέσω τον επόμενο μελητή στο βήμα να σας πω ότι πιθανότερα θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, παρεμβάσεις μετά από τις πρώτες εισηγήσεις και ήδη κ. Μπόγκταν Μπορούσεβιτς, αντιπρόεδρος της ε, Πολωνικής Γερουσίας, ζήτησε τον λόγο εν ώψη αυτής της ζήτησης. Οπότε μπορείτε να προετοιμάσετε και οι υπόλοιποι. Θα έχουμε χρόνο. Οπότε, Ρόζα Μαρία Ρομερό Σάντσες είναι η επόμενη ομιλήτρια από την Ισπανία και έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Για μένα είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Μπορώ να συμμετέχω εξ ονόματος της Ισπανικής Βουλής σε αυτή τη σημαντική δέκατη συνεδρίαση τη κοινοβουλευτική Συντερικής σχέση Ασία Ευρώπη. Κάθε δύο χρόνια αυτή η διάσκεψη μα δίνει την δυνατότητα να μπορέσουμε να ανταλλάσσουμε απόψει για τα θέματα που ε, απασχολούν ε, την παγκόσμια ατζέντα και να παρουσιάσουμε το καθημερινό μας έργο, να μπορέσουμε να βρούμε κοινέ λύσεις σε προβλήματα που συζητάμε σε όλα τα κοινοβούλια και στις χώρες μας και να μπορέσουμε να αναλάβουμε δεσμεύσεις που να βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών μας αλλά και τη λειτουργία των κοινωνιών μας. Η Ευρώπη και η Ασία σήμερα είναι τα δύο μεγαλύτερα οικονομικά μπλοκ του κόσμου και οι εμπορικές ροές που μας ενώνουν ε, είναι ε, οι μεγαλύτερες ε, σε ολόκληρο τον κόσμο. Και φυσικά αυτό θα αυξηθεί στο μέλλον γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ασχολούμαστε και συζητάμε με τη μεταβολή του κλίματος και τις προκλήσεις στον πολυμερισμό. Το θέμα είναι πώς εμείς στις χώρες μας μπορούμε να προωθήσουμε πολιτικές που να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα του παραγωγικού μας συστήματος μέσω πολιτικών και στρατηγικών που να ενισχύουν την βιωσιμότητα των κοινωνιών μας. Θα ήθελα να επικεντρωθώ στην προώθηση της κυκλικής οικονομίας και στο πώς η Ευρώπη και η Ασία μπορούμε να έχουμε ηγετική θέση στη διαδικασία αυτή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αν εφαρμόσουμε την ισχύουσα νομοθεσία για τα πόβλητα, θα δημιουργούνταν πάνω από 400.000 ε, θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις οποίες οι 52.000 θα ήταν στην Ισπανία. Α, ξεκινώ με αυτά τα δεδομένα για να σας δείξω ότι η πρόκληση της κυκλικής οικονομίας ε, θα πρέπει να θεωρείται από όλους ως μια μεγάλη ευκαιρία από την οποία όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε. Η κατάσταση στην Ισπανία που έχει να κάνει με την κατανάλωση πόρων και την ε, τάση των κύριων οικονομικών κλάδων που έχουν ε, επίπτωση στις διαδικασίες κυκλικής οικονομίας θα μπορούσαν να συνοψιστούν μεταξύ τα ε, δεδομένα. Εθνική κατανάλωση υλών στην Ισπανία μειώθηκε περίπου κατά 50% μεταξύ του 2008 και του 2012. Η ε, ενεργειακή ένταση της οικονομίας είναι κατώτερη από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 2013 ήταν η 7η ευρωπαϊκή χώρα με μικρότερη ένταση τα απόβλητα επίσης ε, γενικά ε, μειώνονται στον όγκο τους τα τελευταία χρόνια. Στην περίοδο 2000-2013 η μείωση αυτή ε, σε οικιακά απόβλητα ανακάτοικο έφτασε στο 31,8%. Ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όπου η μείωση ήταν της τάξης του 8%. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ένα φιλόδοξο χάρτη πορείας και να χρησιμοποιήσουμε μια συμμετοχική διαδικασία όπου θα συμμετέχουν ε, όλοι ε, οι παράγοντες και οι πρωταγωνιστές και θα μπορούσαμε να έχουμε και διάφορους στρατηγικούς πρωταγωνιστές σε διάφορα επίπεδα προκειμένου να μπορέσουμε να καθορίσουμε στρατηγικές και φιλόδοξες δράσεις και συντονισμένες δράσεις που να μπορέσουν να εφαρμοστούν με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτός ο χάρτης πορείας, αυτό ο φιλοπορίας θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις κύριες προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας και να συμπεριλαμβάνει κυρίως πολιτικά μέτρα όπως η ανάπτυξη και η εναρμόνιση της νομοθεσίας. Σε αυτό το φόρουμ ε, θέλω να υπογραμμίσω ότι όλα τα διεθνή μέσα που προσυπογράφουν οι νομοθετικές αρχές ε, της Ασίας και της Ευρώπης ε, και έχουν μία διάσταση που αφορά το κλίμα να αποτελέσουν ένα Παράδειγμα, θα πρέπει επίσης να αλλάξουμε το φορολογικό μας σύστημα, να προσφέρουμε κίνητρα που να είναι προσανατολισμένα σε αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο. Τέλος, κυρίες και κύριοι, θέλω να κλείσω απευθύνοντας και μία έκκληση, όπως ήδη έκαναν κάποιοι από τους προλαλήσαντες, μία έκκληση σε όλους και στη σημαντική ευθύνη που έχουμε στα δικά μας κοινοβούλια βάσει τις θέσεις που έχουμε στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας. Οι πολιτικές μας θα πρέπει να προβούν σε μια αλλαγή παραδείγματος, να προωθήσουμε την δημιουργία ενός βιώσιμου οικονομικού μοντέλου, ε, μια διαδικασία που αναμφισβήτητα ε, μπορούν η Ευρώπη και η Ασία να προωθήσουν μέσα από το διάλογο και την συμπληρωματικότητα. εργαστούμε έτσι ώστε το κλίμα συνεργασίας και ανοιχτού πνεύματος μεταξύ των εθνών μας να προωθηθεί. Είμαι πεπισμένη ότι θα θριαμβεύσουμε στην πρόκληση αυτή για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον, ένα καλύτερο πλανήτη όπου οι επόμενες γενιές, τα παιδιά μας θα μπορούσαν να είναι ευτυχισμένοι. Σας ευχαριστώ και καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ροβέρα Σάντσες. Μας είπατε πολλά ενδιαφέροντα σχετικά με τη σημασία της μετατροπής των οικονομιών μας. Ευχαριστώ πολύ που αναφέρεται επίση την κυκλική οικονομία, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα, ο κ. Φουν Κοντσιέν ε, πρόεδρο τη ε, Εθνοσυνόλευση του Βιετνάμ. Παρακαλώ. Κυρία Πρόεδρε, Συμπρόεδρη, επικεφαλής αντιπροσωπιών, κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, μεταβολή του κλίματος, είναι μια μη παραδοσιακή απειλή. Είναι απειλή κατά όλων των χωρών ανεξαιρέτως. Χαίρομαι λοιπόν που σήμερα εδώ συζητούμε το θέμα καθώς και τις συναφείς προκλήσεις για την πολυμερή συνεργασία. Θα συζητήσουμε λοιπόν τις επιπτώσεις της μεταβολής του κλίματος που επηρεάζει τις κυβερνήσεις μας, τον τρόπο διακυβέρνησης την δίμα στην επιβίωση αλλά και απειλεί την πολυμερή συνεργασία. Και τούτο διότι συνεπάγεται συγκρούσεις, χάσματα, ρήγματα, αρχόμενο εθνικισμό, μη παραδοσιακές απειλές κατά της ε, ασφάλειας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει σε πολυμερές επίπεδο όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε. Κυρίε και κύριοι, νομίζω ότι η ΕΣΕΠ μπορεί να είναι υπερήφανη για τη στα θέματα περιβάλλοντος τις τελευταίες δεκαετίες. Καταφέραμε να προωθήσουμε την αϊφορική διαχείριση των φυσικών πόρων. Να συνεχίσουμε λοιπόν στον δρόμο αυτόν τη συνεργασία διότι η μεταβολή του κλίματος έχει επιπτώσεις και στην αυτιλία, στην καθημερινότητα πολλών λαών, στην κοινωνία μας. Ξέρετε το Βιετνάμ είναι μία από τις χώρες που πλήττονται ήδη από την μεταβολή του κλίματος. Για παράδειγμα, δείτε τι γίνεται στον ποταμό Μεκόγκ, που είναι μια εξαιρετικά ευάλωτη περιοχή λόγω της ανόδου της της θάλασσας όπως ε, είναι με τον Γάνγκη στον Μπαγκλαντές ή τον Νίλο στην Αίγυπτο στα αντίστοιχα δέλτα δηλαδή αυτών των ποταμών το κόστος αυτών των επιπτώσεων θα είναι τεράστιο για τον πληθυσμό, για τους ανθρώπους αλλά και τις περιουσίες το Βιετνάμ αναγνωρίζει ότι το φαινόμενο είναι θέμα επιβίωσης είναι όμως και μια ευκαιρία να γίνουμε διεθνώς πιο ανταγωνιστικοί, πιο δυνατοί. Τα τελευταία χρόνια το Βιετνάμ έχει προτείνει και υλοποιήσει διάφορες λύσεις. Είμαστε πλέον μέλος της Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τη Μεταβολή του Κλίματο. Μαζί με άλλε 175 χώρε υπογράψαμε τη Συμφωνία των Παρισίων και συμμετέχουμε στο σχέδιο δράση για την εφαρμογή στην πράξη τη Συμφωνία των Παρισιών. Η Βουλή μας τα τελευταία χρόνια εντείνει τις προσπαθειές της για το περιβάλλον σε πολυμερή φόρα. Για παράδειγμα, συνεργαζόμαστε με την Διακοινοβουλευτική Ένωση. Φιλοξενήσαμε ένα σεμινάριο για τη μεταβολή του κλίματος ειδικά και προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους για το 2020 τους στόχους της εφορικής ανάπτυξης. Επίσης υπερψηφίσαμε απόφαση στο EPPF τον Ιανουάριο του 2018 και κάνουμε ό,τι παίρνει από το χέρι μας για να προωθήσουμε τα θέματα περιβάλλοντος ε, στην 39η Σύνοδο του ΑΣΕΑΝ. Το ΑΣΕΑΝ και το ΑΣΕΠ και η ΑΣΕΠ μάλλον θα μιλήσουν για το κλίμα, θα κάνουν πράγματα για το κλίμα υποβάλλουν συστάσεις και προτάσεις. Έχει πολύ μεγάλη σημασία όμως να ανταλλάξουμε απόψεις και γνώση μεταξύ βουλευτών, ειδικών, μεταξύ επιχειρηματιών για να λάβει ο καθένας την ευθύνη που του αναλογεί. Για να κάνουμε τον κόσμο μας πιο ανθεκτικό. Για να δημιουργήσουμε ευκαιρίες, για να παρακολουθήσουμε την υλοποίηση των διεθνών δεσμεύσεων για το κλίμα να υλοποιήσουμε την ατζέντα για το 2030, το κύριο του πρότοκολ της Συμφωνίας των Παρισίων. Και τρίτον, υποστηρίζουμε την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η την η ΑΣΕΑΝ να δρομολογήσει έναν διάλογο επιθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της ε, ΑΣΕΠ. Εύχομαι στην συνεδρίαση μας κάθε επιτυχία και καλή επιτυχία σε όλους στο έργο σας. Uh, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χέν για τις πολύτιμες αυτές παρατηρήσεις σας. Και τώρα να δώσω το λόγο στον τελευταίο μας προσκεκλημένο ο κύριος Μίσρα από το ε, Εθνικό Κοινοβούλιο της Ινδίας. Κυρίε και κύριοι, εξαιρετούμε πρόεδρε, εξαιρετούμε βουλευτέ. At the outset, let me express my sincere thanks. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα για το γεγονός ότι μου δίνετε την δυνατότητα να μιλήσω εδώ ενώπιον σας σε αυτήν την συνάντησή μας. Είναι μεγάλη μου τιμή. Θέλω να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που φιλοξενεί αυτή τη δέκατη συνάντηση της ΑΣΕΠ και για το γεγονός ότι επέλεξε το θέμα της κλιματικής αλλαγής ένα από τα πλέον πιεστικά και σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στον καιρό μας η ανθρωπότητα. Θέλω μέσα από αυτό το βήμα να σας διαβιβάσω το μήνυμα ότι η Ινδία ε, είναι προσιλωμένη και συνεχίζει τις δεσμεύσεις της για την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει και την αντιμετώπιση των προκλήσεων. ταυτόχρονα με την κοινωνική και οικονομική μας ανάπτυξη δεν χάνουμε από το επίκεντρο της προσοχής μας το περιβάλλον και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με σεβασμό, ισότητα και κλιματική δικαιοσύνη με στόχο να προστατεύσουμε τους φτωχούς και τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες από αυτές τις κλιματικές αλλαγές. Στο πλαίσιο αυτό θέλω να σας αναφέρω ότι οι παροδόσεις μας, η φιλοσοφία μας, οι πρακτικές μας αλλά και οι βιώσιμες καταναλωτικές μας συνήθειες μας βοηθούν στην διατήρηση της φύσης και την αντιμετώπιση των προκλήσεων και γι' αυτό θέλω να σας πω ότι οι παραδοσιακές μας πρακτικές σε συνδυασμό με την σύγχρονη τεχνολογία αντικατοπτρίζονται στα προγράμματα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ανάπτυξης που έχουμε καταρτήσει. Ο πρόεδρος μας, ο, πρωθυπου, ο πρωθυπουργός της χώρας μου, με συγχωρείτε, ο κύριος Ναρέντνα Μόντι, έχει προσδιορίσει τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τα ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή ως εξαιρετικά σημαντικά ύψης της προτεραιότητας για την αλλαγή που θέλουμε να επιφέρουμε στη χώρα μου. Έχει τονίσει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει ε, και λαμβάνει υπόψη του τα συμφέροντα και των μελλοντικών γενεών. Και είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι έχουμε σημειά, σημειώσει μεγάλη πρόοδο στον, στον τομέα του μετριασμού των προβλημάτων περιβαλλοντικής φύσης και στον τομέα της ανάπτυξης περιβαλλοντικών, πολιτικών και τεχνολογιών που θα μας βοηθήσουν στο μέλλον η Συμφωνία των Παρισίων οι πολυμερείς σχέσεις απαιτούν συνεργασία και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Η επιτυχία της συμφωνίας αυτής θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα με την οποία οι χώρες και ιδίως οι αναπτυγμένοι εταίροι μας θα δράσουν ως προς τις δεσμεύσεις τους. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να σας αναφέρω το σχέδιο δράσης του Μπαλί που περιλαμβάνει ένα σημαντικό μηχανισμό για να δοθούν τα εργαλεία και τα μέσα στις αναπτυσσόμενες χώρες προκειμένου και εκείνες να ανταποκριθούν στους περιβαλλοντικούς τους στόχους. Να ενισχύσουν την έρευνα, τη συνεργασία στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Ως αναπτυσσόμενη χώρα, η Ινδία καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή και έχουμε επίγνωση των υποχρεώσεών μας. Είμαστε δεσμευμένοι στο να εξασφαλίσουμε ότι το περιβάλλον και η ανάπτυξη θα συμβαδίσουν, θα πάνε χέρι-χέρι για να επιτύχουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης που έχουμε θέσει. Ο πρωτοπόρος ρόλος της Ινδίας στην ανάπτυξη της ε, παγκόσμιας ηλιακής συμμαχίας έχει λάβει πολύ θετικά σχόλια από ολόκληρο τον κόσμο. Ελπίζω ότι οι συζητήσεις που θα έχουμε σήμερα και αύριο εδώ θα αποδειχθούν γόνιμες και θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των προσπαθειών μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ας σώσουμε λοιπόν τον πλανήτη μας και ας δώσουμε στις μελλοντικές μας γενιές έναν καλύτερο κόσμο.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 Uh, Πρόεδρος, δυστυχώς δεν υπήρχε διερμηνία για τη γλώσσα σας. Σας ευχαριστώ παρόλα αυτά για την τοποθέτησή σας. Λοιπόν, να κάνω κάποιες ανακοινώσεις Προτού περάσουμε στο άτυπο μέρος των συζητήσεων μα. είμαι πολύ χαρούμενη που έχω την ευκαιρία να σας ανακοινώσω ότι πλέον έχουμε οριστικοποιήσει την τελική εκδοχή του κειμένου που θα εγκριθεί αύριο πριν από την καταληκτική συνεδρίασή μας, πριν τις 12 θα εγκριθεί χωρίς συζήτηση γιατί η συζήτηση θα έχει ολοκληρωθεί, η διαδικασία θα έχει ε, ολοκληρωθεί και ε, ε, βρίσκομαι στην πολύ ευχάριστη θέση να σας πω ότι το κείμενο είναι εξαιρετικό. Οι ομιλητές ε, θα μπορούσαν να έχουν δημοσιευμένες τις απόψεις τους στην ιστοσελίδα της ΕΣΕΠ10 αν το επιθυμούν. Επομένως, αν θέλετε, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία και να το φροντίσει και ηλεκτρονικά μπορείτε να τις στείλετε τις ομιλίες σας είτε να τις δώσετε σε χαρτί όπως ε, θέλετε, αλλά νομίζω ότι θα ήταν ε, καλό ε, να διατηρήσουμε έτσι τις εξαιρετικές σας ομιλίες. Mr. Bogdan Borusevich. Θέλω να καλέσω τον κύριο Bogdan Μπορούσεβιτς, τον αντιπρόεδρο του Κοινοβουλίου της Πολωνίας, να πάρει το λόγο. Και μπορείτε να θέσετε ερωτήσεις και να κάνετε σχόλια, αν θέλετε. Μπορείτε να θέσετε ερωτήσει στους ομιλητές μας εδώ στο πάνελ. Ο κ. Μπρούσεβιτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Βρισκόμαστε σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Κανένας δεν είχε αμφισβητήσει τις συμφωνίες των Παρισίων στο παρελθόν τώρα αμφισβητήθηκαν από ένα πολύ σημαντικό κράτος. Δεν ε, συνηθίζαμε να ξανανοίγουμε τη συζήτηση. Όταν ε, όλοι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα κοινό συμφέρον, όμως βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η κατάσταση σήμερα. Βρισκόμαστε σε μια, σε μια διαφορετική κατάσταση. Θα ήθελα να δηλώσω ότι η Πολωνία έχει μειώσει τους, ε, τις εκπομπές διεξιδίου του άνθρακα. τις εκπομπές ορίων του θερμοκηπίου. Είναι τεράστιο επίτευγμα αυτό για την Πολωνία ως χώρα, γιατί η οικονομία μας βασίζεται ε, σε λιγνίτη. Επομένως, είμαστε σε θέση να πρέπει να εξυγχρονίσουμε την οικονομία μας. προκειμένου να τροποποιήσουμε την ε, διαδικασία καύσης λιγνίτη και να επενδύσουμε σε πράσινη ενέργεια. Σε ό,τι αφορά το ενεργειακό μείγμα στην Πολωνία, ο άνθρακας και ο λιγνίτης αυτή τη στιγμή αντιστοιχούν στο 80%. και χρησιμοποιούμε λιγνίτη και άνθρακα κατά 90% στην Πολωνία για την παραγωγή ενέργειας. Όπως ε, και η Φιλανδή πρόεδρος είπε, είδαμε και εμείς κλιματική αλλαγή στην Πολωνία. Έχουμε σαφή αύξηση της θερμοκρασίας μπορούμε να δούμε τις ε, τάσεις τα τελευταία 20-30 χρόνια. Επίσης, έχουμε ακραίες καιρικές συνθήκες στην Πολωνία που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Αυτό σε ευρωπαϊκή κλίμακα, όχι σε ασιατική κλίμακα. Είχαμε τυφώνες, πολύ ισχυρού ανέμους πριν δύο χρόνια. Ο ανέμος κατέστρεψε μεγάλες δασικές εκτάσεις στην Βόρεια Πολωνία. Επομένως, έχουμε βιώσει και εμείς από πρώτο χέρι την κλιματική αλλαγή. Πέρσι, το καλοκαίρι, είχαμε τρομερό καύσιμο στην Πολωνία με θερμοκρασίες που έφταναν τους 30 βαθμούς Κελσίου. Και νομίζαμε ότι βρισκόμασταν στη Μεσόγειο εκείνη την περίοδο. Όλα αυτά καταλήγουν στο εξή. Αν και στο παρελθόν είχαμε κάποιους ανθρώπους που αμφισβητούσαν την αναγκαιότητα μείωση των εκπομπών του άνθρακα, σήμερα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Ανησυχούμε περισσότερο μάλιστα όταν ακούμε κάποιες αναπτυγμένες χώρες να αρχίζουν να αμφισβητούν εκ νέου το θέμα της μεταβολής του κλίματος. Αν ε, ήταν να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση, τότε θα, χάναμε όλα όσα έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα. Και φυσικά δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει το μέλλον σε 20 χρόνια. Σας ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ κύριε Μπορούσεβιτς. Από τις αντιπροσωπείες από την Ασία. Θέλει κανείς το λόγο για να υπάρχει μια εναλλαγή. Γιατί έχω και αιτήματα από την Ευρώπη. Παρακαλώ. Ο κύριος εκεί, πείτε μας. Ποιος είστε. Φιλιππίνες. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι δυνατόν η απόψη μας να είναι μόνο ανάλογη με τις επιπτώσεις που προκαλούμε. Το φαινόμενο είναι πολύ σοβαρό. Δεν θα κάνουμε τίποτα εάν δεν συνεννοηθούμε και αν δεν πετύχουμε συγκεκριμένες συμφωνίες με συγκεκριμένες δράσεις, συγκεκριμένες παρεμβάσεις και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο καθένας στην περιοχή του μικρές ή μεγάλες χώρες προκαλούν επιπτώσεις πολλές φορές, πολλές φορές σοβαρές στο κλίμα. Εμείς ως Φιλιππίνες συμβάλλουμε μόνο σε ποστό 0,3% στις εκπομπές αερίου, των του θερμοκηπίου. Όμως είμαστε σύμφωνα με διάφορες ε, μετρήσεις η πρώτη χώρα που απειλείται από τη μεταβολή του κλίματος γιατί είμαστε εκτεθειμένοι τους ε, παραόντες του κλίματος. Φαίνεται ότι οι εκτιμήσει αυτέ δυστυχώ είναι σωστέ για τι Φιλιππίνες. Τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας συνέβησαν φυσικές καταστροφές αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη βεβαίω ισχύει το ίδιο, χωρίς προηγούμενο. Είχαμε τυφώνες επί 10 ημέρες 10 ε, εκατομμύρια κυβικά μέτρα εδάφου. προκάλεσαν μια τεράστια κατολίσθηση με περίπου χιλιά θύματα. Το 2009 ο τυφώνας Πεπέγ προκάλεσε τεράστιες πλημμύρες στην ίσο Λουζών με 460 περίπου νεκρούς. Την ίδια χρονιά ο τροπικός τυφώνας έπληξε την Μανίλα μετά από καταρακτώδεις βροχές διάρκειας 24 ωρών. 465 θύματα 11 δισεκατομμύρια πέσους ζημιές. Μετά είχαμε άλλες ε, πλημμύρες στο Μιντενάο με 1260 νεκρούς. 2 δισεκατομμύρια πέσους ήταν οι ζημιές. Και ένα χρόνο μόλις μετά ο τυφώνας Παμπλουκίμ κατέστρεψε την ανατολική ακτή του Μιντενάο. Οι ζημίες ανήλθαν σε 37 δισεκατομμύρια πέσους. 1067 ήταν οι νεκροί. Το χειρότερο όμω ήταν ένα χρόνο μετά. Ο υπερτυφώνας Χαγιάν προκάλεσε καταστροφές χωρίς προηγούμενο. Η ζημία ήταν 9 δισεκατομμύρια πέσος, είχαμε πάρα πολλούς εκτοπισμένους και πάνω από 3.600 νεκρούς. Έτσι λοιπόν, περίπου 11.000 άτομα κατέληξαν λόγω αυτών των καταστροφών και όπως σας είπα εμείς συνεισφέρουμε μόνο στο 0,30% των συνολικών εκπομπών σε όλο τον κόσμο αλλά έχουμε υποφέρει από, την καταστροφική, από τον καταστροφικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Ε, Επομένως, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω της ειλικρινούς παγκόσμιας συνεργασίας με συγκεκριμένες τοπικές δράσεις είναι απαραίτητη. Ε, και εδώ αυτό το φόρουμ είναι το καλύτερο φόρουμ προκειμένου να ε, συνομιλήσουμε για τις στρατηγικές και τις ευθύνες μας. Σας ευχαριστούμε που συμμετέχουμε στη διάσκεψη αυτή και δεσμευόμαστε να συνυπογράψουμε την διακήρυξη στην οποία ε, θα φτάσουμε και να εφαρμόσουμε τη διακήρυξη αυτή σε τοπικές δράσεις. Εμείς δεσμευόμαστε για να έχουμε και εγχώριες πολιτικές και δράσεις, ε, κυρίως μέσω δεσμευτικών συμφωνιών όπως η Συμφωνία των Παρισίων θέλουμε να απευθύνουμε κλήσεις στις αναπτυγμένες χώρες να αναλάβουν ηγετική θέση. Επίσης, ε, έχουμε την αύξηση της παγκόσμιας ε, θερμοκρασίας κατά 1,5 ε, βαθμό Κελσίου και προκειμένου εμείς να επιβιώσουμε, αυτό είναι το όριο. Εδώ είναι η αλλαγή του κλίματος, θα πρέπει να προσαρμοστούμε και να μετριάσουμε τον αντίκτυπο της. Είναι ο κοινός μας εχθρός και θα πρέπει να βοηθήσουμε ένα τον άλλο. Thank for Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε αυτές τις τραγικές ε, εμπειρίες μαζί μας. Επόμενος ομιλητής. Μπορώ να πάρω το λόγο. Έχετε κάποια ερώτηση. Γιατί έχω δύο ακόμη άτομα που έχουν ε, δηλώσει. Έχω μια ερώτηση, παρακαλώ. Όταν ε, συζητάμε ένα θέμα όπως η μεταβολή του κλίματος και πώς θα επηρεάσει το μέλλον μας, είπε ο συνάδελφος ότι σε κάποια χρόνια δεν θα είναι βιώσιμος ο πλανήτης. Νομίζω ότι κάθε γραμμάριο και κάθε χιλιόγραμμο που παράγουμε σήμερα καταστρέφει τον πλανήτη. Εμεί έχουμε κάποιους ανθρώπους, παραδείγματο χάρη, ε, που έχουν ε, πάρα πολλά διαμερίσματα, έχουν ε, πολλά, αγαθό, πολλά αγαθά. Αυτά δεν μπορούσαν να συζητηθούν. να δούμε εμείς πώς θα ελέγξουμε αυτή τη διάσταση της μεταβολής του κλίματος. Νομίζω ότι μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε σε κάποιο βαθμό σε αυτό το θέμα. Σας ευχαριστώ. Ίσως θα μπορέσετε να συνεχίσετε αυτό το θέμα και στις παράλληλες συνεδριάσεις σήμερα το απόγευμα. Να αναφέρω ότι έχουμε αντιπροσωπεία από το βουλή της, από το Κογκρέσο της Ινδίας και ουσιαστικά υλοποιούν μία επίσκεψη μία εβδομάδας για να έρθουν και να γνωρίσουν το έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίως της διοίκησης. Από ό,τι μου ενημέρωσαν, πρόκειται για μία ετήσια παράδοση. Σας καλωσορίζουμε εδώ. Είναι πολύ θετικό το ότι βρίσκεστε εδώ. Δύο άτομα έχουν ζητήσει το λόγο. Και στη συνέχεια δεν νομίζω ότι έχουμε περισσότερο χρόνο ο κύριος Τσαμπολίλο από τη Γερουσία της Ιταλίας να πάρει το λόγο. Και θα σας ζητούσα να μην μιλήσετε παραπάνω από δύο λεπτά, γιατί πρέπει στη συνέχεια να βγάλουμε την οικογενειακή φωτογραφία και να διακόψουμε για το γεύμα. Ευχαριστώ. Λέγομαι Λέλο Τσαμπολίνο. Καλημέρα σε όλους. Πολύ συχνά ξεχνάμε ότι η κύρια αιτία της ε, παγκόσμιας ρήπανσης αλλά και της μεταβολής του κλίματος ε, είναι ακριβώς η κτηνοτροφία. Πολύ συχνά μιλάμε για την κτηνοτροφία, για παραγωγή κρέατος και για την παραγωγή γάλακτος. Και φυσικά και όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Εγώ αντιμετωπίζω πολύ θετικά όλα αυτά που μας ε, ανέφερε εκείνο, όλα αυτά τα θετικά νούμερα. Όμως, ε, αλλά και στην Κίνα, αλλά και σε όλο τον πλανήτη έχουμε πάνω από 700.000 χείρους που εκτρέφονται και αυτό αντιστοιχεί στο 50% της κτηνοτροφίας ε, χείρων παγκοσμίων. Αυτό ε, ουσιαστικά οδηγεί στην ε, δημιουργία πολλών εκπομπών και μιλάμε για πάνω από 30 δισεκατομμύρια τόνους διοξιδίου του άνθρακα και οι μισές από αυτές τις εκπομπές προέρχονται από την κτηνοτροφία. Και η Greenpeace έχει παρέμβει επί του θέματος και μας είπε ότι η κτηνοτροφία μπορεί να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην υγεία και μιλάμε κυρίως για την ε, αντίσταση στα αντιβιωτικά. Έτσι λοιπόν, ίσως ε, θα έπρεπε να προτείνουμε να έχουμε βιώσιμη κτηνοτροφία αλλά και να μην παρέχουμε ε, πλέον επιδοτήσεις για την κτηνοτροφία γιατί παράγουν ε, άζωτο, φόσφορο, ε, αμμονία και επίσης έχουμε και διάφορα σωματίδια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η ΕΦΣΑ, το ECDC, που είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη των Νόσων, δήλωσαν ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές στην υγεία. Και θέλω να κλείσω με μια παράθεση του καθηγητή Peter Spitz από το Μπερντίν στη Σκωτία, που είπε η αναγκαιότητα να μειώσουμε την ε, ζήτηση και την ε, ε κατανάλωση της ε, κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών είναι κάτι επίγον. Μόνο αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα κατάλληλο σύστημα παραγωγής κτηνοτροφίας στο μέλλον θα μας οδηγήσει σε μια βιώσιμη κατάσταση. Βέβαια, ε, εγώ θα έλεγα ότι ε, ακόμη και αν δεν τρώμε καθόλου κρέας, αυτό βελτιώνει την υγεία μας. Αν γίνει κάτι τέτοιο λοιπόν, θα έχουμε μια σημαντική μείωση της ρήπανσης και μάλιστα θα εγγυθεί in primis την ευημερία των ζώων, την ε, ευημερία του ανθρώπου, αλλά θα εγγυθεί και μια καλύτερη υγεία για τον πλανήτη. Ευχαριστώ πολύ. Επιβεβαιώνω ότι πρόκειται για μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει, στην Ευρώπη τουλάχιστον, ότι σε πλανητικό επίπεδο χρειάζεται να υπάρξει μια σταδιακή μείωση της υπερβολικής τουλάχιστον χρήσης ε, ζωικών προϊόντων. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Άραμ Γκάβερ, ε, κεφαλής πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος του Πολωνικού Κοινοβουλίου. Μπορείτε, σας παρακαλώ, όσο πιο σύντομα μπορείτε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να τονίσω τη σημασία που έχει η σημερινή μας συζήτηση και, τον, ε, και τα ζητήματα που συζητούμε, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Τα αποτελέσματα των συμφωνιών του Παρισιού αποτέλεσαν μια εθελοντική μέθοδο επίτευξης των στόχων της συμφωνίας και αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την επίτευξη των στόχων αυτό για την μείωση των εκπομπών και της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Η η Πολωνία ε, έχει επιτύχει ήδη εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έχουμε μειώσει τις εκπομπές μας κατά 30% περίπου ήδη, ενώ ο στόχος υπό το Κιώτο ήταν 6%. Νομίζω ότι μπορούμε λοιπόν να είμαστε περήφανοι για τα όσα έχουμε επιτύχει. Παρόλα αυτά, ε, λόγω της οικονομίας μας, των τεχνολογιών μας και των φυσικών μας πόρων, υπάρχει περαιτέρω περιθώριο μείωσης των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι τα ορυκτά καύσιμα ε, σχετίζονται και με την ενεργειακή μας ασφάλεια. Ακολουθούμε λοιπόν την πορεία μείωσης των εκπομπών με έναν τρόπο που δεν θα πλήξει την ενεργειακή μας ασφάλεια. Η οικονομία μας εξαρτάται από τα ορυκτά καύσιμα μεν, ωστόσο Όλο ένα και περισσότερο εισάγουμε μοντέρνες τεχνολογίες χρησιμοποιώντας την υδροελεκτρική ενέργεια, αιωλική ενέργεια και άλλες τεχνολογίες που μας δίνουν τη δυνατότητα να επιτυγχάνουμε ολοένα και καλύτερα ε, αποτελέσματα υπό τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν βεβαίως στη χώρα μου. Επίσης έχουμε θεσπίσει νόμο για την καθαρότητα του αέρα στην Πολωνία βάσει του οποίου θα ξοδέψουμε τα επόμενα 10 χρόνια 25 δισεκατομμύρια ευρώ για την προστασία της ποιότητας του αέρα και για την καλύτερη διαχείριση της παραγωγής ενέργειας. Η συνεργασία λοιπόν είναι πολύ σημαντική στα ζητήματα που σχετίζονται με το κλίμα. Χρειάζεται συνεργασία συμπράξεις συνέργειας για να αξιοποιήσουμε όλες τις δυνατότητες και τεχνολογίες που έχουμε πλέον στα χέρια μας. Όμως πρέπει να υπάρχει και αλληλεγγύη και δίκαιοι κανόνες για όλους. Και αυτό παρό το γεγονός ότι δεν είναι το βασικό μας θέμα στη στο σημερινή μας συνάντηση πρέπει να σας πω ότι στο ευρωπαϊκό επίπεδο ο Nord Stream είναι ένα τουλάχιστον αμφιλεγόμενο project γιατί ακριβώς δεν συνδέεται ή δεν διαπνέεται από αυτό το πνεύμα αλληλεγγύης που θεωρώ ότι ε, είναι αναγκαίο. Σας προσκαλώ με την ευκαιρία της τοποθέτησής μου βεβαίως και στο Κατοβίτσα όπου θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε βάθος τα ζητήματα που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, και νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ε, συζήτηση αυτή. Νομίζω ότι η συζήτησή μας επικεντρώθηκε ε, σε αυτά που είχαμε συμφωνήσει ότι θα ήταν τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σε αυτή την ΑΣΕΠ 10. Έχουμε λοιπόν ακούσει πολύ σημαντικές παρεμβάσεις που θα τροφοδοτήσουν τις συζητήσεις που θα γίνουν στις, στα θεματικά πάνελ που θα ξεκινήσουν στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ για τη ζωηρή αυτή συζήτηση. Ε, ελπίζω και φαντάζομαι ότι θα σας δω και στις ομάδες εργασίας του απογεύματος και θα πρότεινα τώρα να βγάλουμε την οικογενειακή φωτογραφία, την παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία, να κατεβούμε εμείς όσοι είμαστε στο βήμα κάτω και αν μπορείτε όλοι εσείς που είστε εδώ στην αίθουσα να έρθετε λίγο πιο πολύ εδώ στις πρώτες σειρές στο κέντρο μετά στη μία ε, θα έχουμε το γεύμα μας στην αίθουσα Γεχούντι Μενουχίν που είναι στον πρώτο όροφο του κτηρίου στο οποίο βρισκόμαστε και μετά σας παρακαλώ να προσέλθετε όπως έχει προγραμματιστεί στις 3 ώρες ώρα στις θεματικές μας συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ.